και κυρίως από ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας της. Και είναι σημαντικό που είχαμε και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου που αναφέρεται στα αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα που έπληξαν την Ευρώπη τον προηγούμενο αιώνα και παραμένουν ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας μας. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος οδήγησε σε ανήκουστα επίπεδα ε, βλάβης του κόσμου. Τόσοι υπέφεραν εκατομμύρια ε, βασανίστηκαν, δολοφονήθηκαν, αναγκάστηκαν ε, ε, να πάνε αλλού. Είναι η φρίκη του πολέμου που έπληξε την Ευρώπη και κανείς δεν πρέπει να τα ξεχνάει όλα αυτά. Και γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε τις κοινέ μας αξίες και τις γενικές αρχές πάνω στις οποίες δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σεβόμαστε την ανθρώπινη εξωπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου, και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευτυχώ, οι περισσότερες από τις νέες γενιές στην Ευρώπη δεν υπέφεραν από ολοκληρωτικά καθεστώτα. Όμως, υπάρχει ο κίνδυνος αυτές τις κοινέ αξίες και τις αρχέ να τις θεωρούμε δεδομένες το τραγικό παρελθόν της Ευρώπης πρέπει να χρησιμεύσει σαν ε, ηθικό κίνητρο για να αντιμετωπίσουμε το σημερινό κόσμο. Οι κοινές αξίες που επέτρεψαν να έχουμε τόσα πολλά χρόνια ειρήνη στην Ευρώπη πρέπει να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο των δημοκρατικών μας κοινωνιών και πρέπει να προστατευτούν και ε, να προστατευτούν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι μας δίδαξαν να μην επικεντρωνόμαστε στις διαφορές μας, αλλά ε, σε αυτά που μας ενώνουν. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν ε, μάθει γενιά μετά από γενιά τι σημαίνει η συμμετοχή στην κοινωνία, τι σημαίνει η ανοχή. Παρά τις θετικές εξελίξεις ε, που έχουμε στην Ευρώπη, παρόλα αυτά η Ευρώπη έχει περάσει από πολέμους και από καταστροφές και τη δεκαετία του 90. Και στη δικιά μου χώρα, για παράδειγμα, που η εμπειρία αυτού του πολέμου παραμένει στις μνήμες μας. Αλλά αυτό είναι ένας παραπάνω λόγος για να σεβαστούμε όλη την ειρήνη, την ασφάλεια που προσφέρει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και ενώ πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε τα επιτεύγματα αυτά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σήμερα οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις. Έχουμε την ξενοφοβία, τον εθνικισμό, τον λαϊκισμό, ε, βία, ριζοσπιστικοποίηση Είναι μερικά μόνο από αυτά τα φαινόμενα. Περίπλοκα φαινόμενα τα οποία δύσκολα αντιμετωπίζονται και δεν υπάρχει καμία εύκολη λύση. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι προσεκτική και να αντιμετωπίζει και να καταπολεμάει την προπαγάνδα που μιλάει για εύκολε λύσει. Αυτέ οι υποσχέσει ποτέ δεν μπορεί να υλοποιηθούν. Προσπαθούν να διχάσουν τις κοινωνίες μας, να πούν ότι είμαστε εμείς και εκείνοι, φίλοι και εχθροί. Κάτι το οποίο υπονομεύει όμως τη δημοκρατική και την πολιτικά ανοιχτή συζήτηση. Ο εξτρεμισμός κερδίζει έδαφος. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες για να αποφύγουμε την αδιαλαξία και την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Ε, πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, θέλω να τελειώσω τονίζοντα ότι πρέπει όλοι να θυμόμαστε την ιστορία μα και να μαθαίνουμε από το παρελθόν. Να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη για τα οποία ίσως να είμαστε υπεύθυνοι. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ το Συμβούλιο για αυτή την ομιλία. Συνεχίζουμε με την κυρία Γιώργο από την Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή τη συζήτηση, η συλλογική μας ιστορία και το πώς την απομνημονεύουμε και την μνημονεύουμε και την ε, παρουσιάζουμε είναι σημαντική για το παρόν και για το μέλλον της Ευρώπης. Όπως ε, λέει η φημισμένη ρίση, όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν τη δική τους άποψη, αλλά όχι να διαστρεβλώνουν τα γεγονότα. Και ρόλος της Κομισιόν εδώ είναι να μιλάει για τα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει κάθετα οποιασδήποτε ισχυρισμού, ψευδεί ισχυρισμού που προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ή να παρουσιάσουν τα θύματα όπως την Πολωνία ως εγκληματίες. Δεν θα ανεχθεί η Επιτροπή τέτοιες επιθέσεις κατά της Πολωνίας και παραμένει αλληλέγγυα με την Πολωνία και τον πολωνικό λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπίδησε, αναγεννήθηκε από τις τάχτες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος και μέσα στον ε, ψυχρό πόλεμο αυτές οι αρχές χρησιμοποιήθηκαν για να οικοδομήσουμε ένα κοινό μέλλον. Δεν μπορούμε να συζητάμε τέτοια ιστορικά γεγονότα. Το σύμφωνο Χίτλερ και Στάλιν που υπογράφηκε μεταξύ τους Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης στις 23 Αυγούστου του 1939 άνοιξε το δρόμο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η συμμαχία Ναζί και Σοβιετικής Ένωσης ε, άνοιξε το δρόμο για τον πόλεμο στις 7 Σεπτεμβρίου του 1939 και μετά την είσοδο ε, για τις σοβιετικά στρατεύματα στις 20 ε, Σεπτεμβρίου. Αυτά τα γεγονότα σημάδεψαν την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά είναι τα γεγονότα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την κατάληψη των χωρών της Βαλτικής και της Βεσαραβίας χωρίστηκε η Ήπειρος σε περιοχές επιρροής ε, κακόβουλων καθεστώτων. Πρέπει να επισημάνουμε τις φρίκες που διέπραξαν και τα δύο καθεστώτα. Το οργανωμένο, η οργανωμένη γενοκτονία της, ε, ε της ε, ναζιστικής Γερμανίας ε, τις ζωές εκατομμυρίων ε, Εβραίων, Πολωνών, Ρωμά και άλλων εθνικοτήτων. Ναι, η ιστορία είναι κάτι περίπλοκο. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε το ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης των Σοβιετών στρατοετών σε κρίσιμες στιγμές του πολέμου όταν ο Στάλιν και ο Χίτλερ έγιναν εχθροί. Οι Σοβιετικοί στρατιώτες ήταν οι πρώτοι που έδιωξαν τους Γερμανούς ε, στρατιώτες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μετά από τεράστιες θυσίες από τους λαούς της Σοβιετικής, Ευρώπης, της Σοβιετικής Ένωσης. Έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση ε, στο Auschwitz του Μπέργεναου των στρατοπέδων συγκέντρωσης στην ε, Πολωνία. Στις 27 Ιανουαρίου θα μνημονεύσουμε τα γεγονότα αυτά. Ακόμη και μετά τον πόλεμο, πολλοί άνθρωποι από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη συνέχισαν για δεκαετίες να υποφέρουν υπό το απολυταρχικό καθεστώς των κομμουνιστικών καθεστώτων. Καθεστώτα τα οποία συχνά εγκαθιδρύθηκαν με την υποστήριξη και κατά τη βούληση των τοπικών πληθυσμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε στις 23, της 23 Αυγούστου ως επίσημη ημέρα μνημονευσής των εκατομμυρίων θυμάτων των απολυταρχικών καθεστώτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να συμβάλλει μαζί με την ευθύνη της για την προώθηση της ε, μνήμη ε, των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει από λιταρχικά καθεστώτα στην Ευρώπη και η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εορτάζουν και αυτά αυτή την πανευρωπαϊκή Μέρα μνημόνευσης αυτών των ιστορικών γεγονότων. Είναι καθήκον μας να θυμόμαστε τα ονόματα των εκατομμύριων που διώχθηκαν και να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους. Και επίσης να μελετάμε επιμελώς τους κανόνες, τους λόγους ε, και τη συμπεριφορά των απολυταρχικών καθεστώτων. Ειδικότερα διότι σήμερα, 81 χρόνια μετά από το άνοιγμα αυτού του σκοτεινού κεφαλαίου στην ευρωπαϊκή ιστορία, οι κοινέ μα αξίε, ε, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτο δικαίου και η δημοκρατία ε, βρίσκονται πάλι υπό απειλή από εξτρεμιστέ, εθνικιστέ και από ε, ρητορική που διχάζει τον κόσμο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτά τα γεγονότα για να καταλάβουμε τη δική μας ιστορία και να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Το όνειρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σχηματίστηκε αμέσως μετά τον πόλεμο με σαφή στόχο τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού θεμελίου για μακροχρόνια ειρήνη στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρώπη να είναι απόλυτα σαφής για τα θέματα αυτά. Η διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων αποτελεί απειλή για τις δημοκρατικές μας κοινωνίες και θα πρέπει να καταπολεμηθεί όπου αυτό είναι δυνατόν. Η οργανωμένη και στοχευμένη διάδοση διαστρεβλώσεων και παραπληροφόρησης είναι κάτι που θα πρέπει να μας βρίσκει αντίθετος. Θα πρέπει να την απορρίπτουμε και εγώ η ίδια θα καταβάλω προσπάθειες υπό το δικό μου αξίωμα να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία να μας επιτρέψει να ε, απελευθερωθούμε από αυτές τις απειλές. Αξιότιμα μελή, κυρίες και κύριοι, αναμένω με ανυπομονησία τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Γιούροβα, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα οι πολιτικέ ομάδε. Πρώτα, πρώτα η Σάντρα Καλνιέτα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ. κύριε Επίτροπε, να σας τα πω στην μητρική μου γλώσσα, τα λεδονικά. Βάλτε τα ακουστικά σας. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, γιορτάζουμε 70 χρόνια από την νίκη των συμμάχων. Είπα, Βρετανία, Γαλλία και Σοβιτική Ένωση. Μας αρέσει να λέμε ότι νικήσαμε. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Το 1939 υπήρξε αυτή η συμφωνία για την διαίρεση της Ευρώπης, το, το, το, το μοίρασμα, τη μοιρασιά μεταξύ Χίτλερ και Στάλιν. Οπότε επιτέθηκε στην ε, Πολωνία ε, ο Χίτλερ ε, μετά τη συμφωνία και έμεινε μόνο η Βρετανία να υπερασπίσει την Ευρώπη και μιλούμε για το Σεπτέμβριο του 1939 μέχρι τον Ιούνιο του 1941. Οπότε ο Στάλιν μέχρι τότε όλη αυτή την περίοδο ήταν σύμμαχος του Χίτλερ. Επομένως η Σοβιετική Ένωση είναι συνυπεύθυνη. Συνυπεύθυνη του ξεκινήματος του πολέμου. Αυτό δεν σβήνεται με τίποτα. Ούτε καν με όλες αυτές τις προσπάθειες αλλίωσης της ε, ιστορίας. Βεβαίως υπήρξε ηρωισμός από πλευράς του λαού, υπήρξαν τεράστιες θυσίες από πλευράς του σοβιετικού λαού. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Πρέπει να τα θυμόμαστε για πάντα, λέει η κυρία Καλνιέτα, πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καλνιέτε. Επόμενος ομιλητής από τους Σοσιαλδημοκράτες, ο κύριος Γκάγερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδέλφοι. Κυρία Γιούροβα, συμφωνώ. Κανείς δεν μπορεί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα. Μετά από όσα ακούσουμε, θα θέλω να υπογραμμίσω διπλά αυτό που είπατε. Θα πρέπει να σας θυμίσω γιατί καθόμαστε εδώ. Η αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή της συνεργασίας των ευρωπαϊκών λαών ήταν το προήμιο το οποίο μας θυμίζει ότι η αρχική μας συνθήκη δεν ήταν παρά ε, μια αρχική συμφωνία για τον άνθρακα και το χάλιβα αλλά με την πεποίθηση ότι πρέπει να εμπορευόμαστε μεταξύ μας, να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας ε, και ότι χρειαζόμαστε κοινού θεσμούς ε, που να προωθούν την ειρήνη. Το πόσο επιτυχές είναι αυτό το μοντέλο το βλέπουμε σήμερα, ότι σήμερα δεν μιλάμε πια για άνθρακα και χάλιβα μόνο, αλλά για πολλά άλλα Χρειαζόμαστε στην Ευρώπη να μιλάμε ανοιχτά. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση τη δημοσιογραφίας. Ε, δεν πρέπει να αφήνουμε να απειλούνται οι δημοσιογράφοι. Θέλουμε να υπάρχει ελεύθερο ραδιόφωνο, δεν πρέπει να το αφήνουμε να τίθεται υπό απειλή στα κράτη-μέλη. Ω εμεί, ε, ε, ω αιρετοί πολιτικοί, πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκάιερ. Τώρα εκ μέρους του Renew, ο κύριος Σάρλς Γκέρνς έχει το λόγο. Παρακαλώ. Η διαχείριση του παρελθόντος είναι λεπτή υπόθεση και φαίνεται λεπτή, είναι δύσκολη, αλλά είναι και αναγκαία. Και νομίζω ότι ο Ζαν Κάν ο οποίος ξεκίνησε το παρατηρητήριο της Ευρώπης για το ρατσισμό και την ξενοφωνία, κάτι θα μπορούσε να μας πει γι' αυτό. Δυστυχώς μας εγκατέλειψε. Ε, θα έπρεπε να καταγραφούν όλες αυτές οι ενωσίες που κατά παράλογα ε, και να υπάρχουν στα βιβλία της ιστορίας. Και ένα από τα πιο παράλογα πράγματα που έχουμε συναντήσει είναι κάτι σε ιστορικό βιβλίο της Αυστρίας ότι ήταν το πρώτο θύμα του Τρίτου Ράιχ. Να, τι συμβαίνει όταν δεν μεταχειριζόμαστε τα θέματα του παρελθόντος όπως πρέπει, όταν δεν έχουμε το θάρρος να τα εξετάσουμε. Και είναι πράγματι πολλοί αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην παραπληροφόρηση. Αυτοί οι οποίοι διαστρεβλώνουν την ιστορική πραγματικότητα, είτε αγνώντας τα διαφυσβήτητα ιστορικά στοιχεία, είτε αρνούνται να τα χρησιμοποιήσουν σαν σημείο αναφοράς. Η δεύτερη περίπτωση είναι μάλιστα χειρότερη από την πρώτη. Γιατί την ανοησία, άντε εντάξει, κανεί μπορεί να πει ότι δικαιολογείται κάτω από κάποιε συνθήκε. Αλλά το δεύτερο, όχι. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε απέναντι σε αυτούς τους αρνητές της ιστορίας. Πώς μπορούμε να αντιταθούμε σε αυτούς που δολοφονούν τη μνήμη, όπως τους λέει και ο Βινταλακέ. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε, πιστεύω, που βέβαια δεν θα υλοποιηθεί αμέσω, αλλά όπως οι μάρτυρες, ε, καθώς ε, όσοι έζησαν αυτά τα γεγονότα ε, μας έχουν εγκαταλείψει, θα έπρεπε να ξαναδούμε τα χέρια της ιστορίας. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα, από το οποίο πρέπει να εμπνευστούμε. Η Γερμανική Ομοσπονδία στην έκδοση της Bundesland πριν αντιμετώπισε το παρελθόν της, είχε το θάρρος να το κάνει. Και με θάρρος λοιπόν αντιμετώπισε το παρελθόν της χωρίς να κρύψει τίποτα και στα ιστορικά εγχειρίδια αλλά και στα μέσα ενημέρωσης φρόντισε για την αλήθεια. Και τα νέα, ε, στα νέα γερμανικά κρατήδια όμως δεν έγινε αυτό. Οι προσπάθειες που έγιναν για να μάθει κανείς την ιστορία και για να μαθαίνει την ιστορία ποτέ δεν είναι μάτες. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρενς. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους των Πρασίνων και της Ελεύθερης Συμμαχίας, ο κύριος Μπετικόφερ. Παρακαλώ κύριε Μπετικόφερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Γιούροβα, σας ευχαριστώ πολύ που φέρατε την Πολωνία σε αυτή την συζήτηση και πάλι. Πρόσφατα είχαμε όλο και περισσότερες συζητήσεις για την ιστορία και δεν είναι εύκολο κανείς να συζητά για τέτοια θέματα. Δεν είναι ο ρόλος μας, η ευθύνη μας να αθώσουμε οποιονδήποτε από οποιοδήποτε ιστορικό γεγονός. Και την ιστορική αλήθεια δεν την έχει κανείς στη διάθεσή του ούτε καν κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Όμως πρέπει να υποστηρίζουμε τα γεγονότα όπως καλύτερα τα γνωρίζουμε αυτά. Και αυτό έχει να κάνει με τη Σοβιετική επίθεση, αυτό έχει να κάνει με ό,τι έχουν υποφέρει οι Σοβιετικοί, αλλά έχει να κάνει και με τον ρόλο που έπαιξαν ε, οι διάφοροι που φρόντισαν για την ειρήνη στη συνέχεια. Και όταν ένα θύμα γίνεται ο θήτης ενός εγκλήματος, επίσης πρέπει να υψώνουμε τη φωνή μας. Και αν κάποιος λύκος φωνάζει «Α, λύκος», και αυτό πρέπει να το καταγγείλουμε. Τέτοιου είδους ε, συζητήσεις όμως σπάνια αφορούν μόνο το παρελθόν. Το να μεταφέρουμε τις καταγγελίες από τον ένα στον άλλον οδηγεί στο να καταλήγουμε σε έναν στόχο και μάλιστα όχι μόνο για μία επίθεση. Αυτό πρέπει να το προσέξει η Ευρώπη. Εγώ και Ευχαριστούμε κύριε Μπιουτικόφερ για την ομάδα ID ο Αλισάνδρο Πάντσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δυστυχώς είναι πολλές οι διαστρεβλώσεις που ακούμε για ιστορικά θέματα και για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη. Η αντίσταση στην Ιταλία είναι αναπόφευκτο θέμα, αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Αντιθέτως, δεν θέλω να δαιμονοποιούμε κάποιους. Απλά θέλω να κάνω κάποιε διευκρινήσει στην Ιταλία. Δεν υπήρχε μόνο μία ομάδα παρτιζάνων που μαχήθηκε κατά των φασιστών. Υπήρξαν κομμουνιστέ, σοσιαλιστέ, καθολικοί, συντηρητικοί και ρεπουμπλικάνοι. Παρ' όλα αυτά στη χώρα μου το αφήγημα ε, είναι διαστρεβλωμένο. Αυτό στο οποίο μόνο κάποιοι μαχήθηκαν κατά του φασισμού και υπό αυτό το φως ορισμένες ενώσεις ε, λαμβάνουν και δημόσια χρήματα και αντί να εξηγούν αντικειμενικά την ιστορία δεν χάνουν καμία ευκαιρία για να ξεχωρίσουν πολιτικά και να σταθούν μαζί με την ε, αριστερά στην Ιταλία κατά τον ε, εμφύλιο πόλεμο 43-45 εγκλήματα έκαναν και οι δύο πλευρές. Ωστόσο για τα εγκλήματα των φασιστών τα ε, περιγράφουμε μια χαρά. Τα εγκλήματα των παρτιζάνων σαν να υπάρχει ατιμορρησία, να τα έχουμε ξεχάσει. Ας δούμε την ιστορία του Λοραντορίντιο, ε, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους παρτιζάνους. Πάνω από 2.600 γυναίκες βιάστηκαν και σκοτώθηκαν χωρίς ε, δίκη με την αιτιολογία ότι ήταν φίλες με τους φασίστες. Ωραία είναι να κρυβόμαστε πίσω από τραγούδια όπως τον Μπελατσάο, όπως κάνουν κάποιοι επίτροποι εδώ. Ενώ γνωρίζουμε αντιθέτως ε, ότι το Μπελατσάο δεν ήταν ύμνος των Παρτιζάνων. Θέλω να αναφέρω ένα μεγάλο δημοσιογράφο τη αριστερά που χάσαμε πριν λίγε μέρε. Όλοι τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, τα έχουν ακούσει. Κανεί δεν τολμά να τα πει δημοσίω γιατί φοβάται να τον χαρακτηρίσουν φασίστα. Ευχαριστώ για την ε, πνευματική σας ειλικρίνεια, Τζαν Παύλο Πάντσα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάντσα. Μία μικρή υπενθύμηση. Πρέπει να τηρείτε το χρόνο αγόρευσης που σας έχουμε δώσει. Και σας υπενθυμίζω δεν υπάρχει μπλε κάρτα. Και δεν μπορείτε να ε, ζητήσετε να παρέμβετε τώρα Έχουμε ήδη τον κατάλογο. Αυτό σα υπενθυμίζω δεδομένων των συζητήσεων που έχουμε να κάνουμε για την επικαιρότητα. Α περάσουμε στην επόμενη παρέμβαση εκ μέρου των ECR, η κυρία Φωτίγκα. Αγαπητοί συνάδελφοι, από σας ευχαριστώ όλους σας που υιοθετήσατε αυτό το ψήφισμα του Σεπτεμβρίου για την κοινή μνημόνευση που βασίζεται σε ισόρροπα στοιχεία και σε γεγονότα. Από την αρχή και τα δύο μέρη της συμφωνίας Χίτλερ και Στάλιν χρησιμοποίησαν ε, ψέματα, ε, εκτρετής αμαύρωσης ε, και, ψέμ και απάτες για να κάνουν αυτό που ήθελαν με το ολοκαύτωμα. Ο Χίτλερ κατηγόρησε τους Εβραίους για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μήνες μετά από τη διάπραξη του εγκλήματος πολέμου σε πάνω από 20.000 πολωνικά μέλη ε, στο Κατίν και σε άλλα μέρη ο Στάλιν ενημέρωσε τους ε, Πολωνούς στρατηγούς 20 και τους λοιπούς ότι τους ε, απελευθέρωσαν και ότι ξέφυγαν αυτοί και πήγαν στη Μαντζουρία αργότερα κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στο Πότσνταμ διαπράχθηκε ένα άλλο έγκλημα πολέμου κατά Πολωνών και Λιθουανών. Αυτό ονομάστηκε η συγκέντρωση του Αυγούστου. Δυστυχώς σε αυτή τη διαδικασία μαύρωσης κατηγορείται η Πολωνία και άλλες ε, χώρες και έτσι ο πρόεδρος Πούτιν χρησιμοποιεί τους ίδιους μύθους. όπως χρησιμοποίησαν τότε και τα δύο μέρη της συμφωνίας Χίτλερ και Στάλιν. επιπλέον δοξάζει τον Στάλιν και τις δραστηριότητές του και σε λαμβάνει υπόψη για τις σημερινές του πολιτικές. Θα πρέπει να το θέσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φωτίγκα για την QNGL ή κυρία Κατερίνα Κονέτσνα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν μια μεγάλη καταστροφή. Είχαμε την καταρρεύση των χρηματιστηρίων, οικονομικό χτύπημα προς όλο τον κόσμο, φτώχεια και πείνα για εκατομμύρια ό,τι ακουγόταν που τους έδινε ελπίδα αρπαζόντουσαν από αυτό. Έτσι έγινε και με τον ναζισμό και με τον φασισμό. Ε, Βερολίνο, Ισπανία, ε, Ιταλία. Έτσι έγινε με αυτούς τους δικτάτορες. Η Τσεχοσλοβακία προδόθηκε από τους συμμάχους της στο Μόναχο. Η Ευρώπη απέτυχε γιατί έβλεπε αδρανός να παραβιάζονται όλες οι συμφωνίες. Έμεινε απροστάτευτη η Τσεχοσλοβακία. Άουσβιτς, Νταχάου, εκατομμύρια νεκρών. Ε, χτυπήθηκε, διαλύθηκε όλη η Ήπειρος. Θα πρέπει να δείξουμε σεβασμό στους νεκρούς και όσοι εγκλημάτισαν θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι στιγματισμένοι και να τιμούμε τους απελευθερωτές η πρόεδρος. Και τώρα. Το λόγο έχει ο κύριος Νικολάου Αλαβάνος ε, από τους μη γεγραμμένους. Έχετε το λόγο. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία σας. Γιατί παρά τις αντικομουνιστικές αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, την εκστρατεία ψέματος, διαστρέβλωσης της ιστορίας, την προκλητική εξίσωση του κομμουνισμού με το τέρας του φασισμού, τα δισεκατομμύρια ευρώ για προγράμματα φρονηματισμού της νεολαίας δεν έχετε καταφέρει να ξαναγράψετε την ιστορία. γι' αυτό για μήνες κρατάτε την αντικομουνιστική μηχανή σε ψηλές τροφές με το κατάπτυστο αντικομουνιστικό ψήφισμα του σεπτεμβρίου με αλλεπάλληλες συζητήσεις αντικομουνιστικού χαρακτήρα σε κάθε ολομέλεια. ο αντικομουνισμός είναι στο dna της ευρωπαϊκής ένωσης και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής οι λαοί το ξέρουν το βλέπουν αποθράσινση φασιστικών και εγκληματικών ομάδων ανάμεσά τους και η υπόδικη ναζιστική χρυσή αυγή στην ελλάδα απαγορεύσεις κομμουνιστικών κομμάτων σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης στην πολωνία στις χώρες της βαλτικής περιορίζοντας τη δράση των κομμουνιστών περιορίζοντας τη συμμετοχή τους στις εκλογές με διώξεις αγωνιστών με ξύλωμα ιστορικών μνημείων. δεν θα τα καταφέρετε όσο και αν πασχίζετε να βαφτίσετε τη μέρα της αντιφασιστικής νίκης. σε μέρα της ευρώπης η αλήθεια θα λάμψει γιατί φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια από το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου τότε που το χιτλεροφασισμό τον τσάκισε υπάλληλοι των λαών με επικεφαλής τους κομμουνιστές τη σοβιετική ένωση και τον κόκκινο στρατό. το μέλλον των λαών δεν συμβιβάζεται με την καπιταλιστική εκμετάλλευση με τη φτώχεια τον πόλεμο και την προσφυγιά. ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον. Κύριε Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Νικολάου Αλαβάνο και τώρα θα δώσουμε το λόγο στου συναδέλφου πρώτα από τον Αντρέα Χαλίσκη που έχει ένα λεπτό. Εγώ έρχομαι από την Πολωνία. Είμαι ένας εξ αυτών που ανέλαβε την πρωτοβουλία για αυτή την συζήτηση και ευχαριστώ το Σώμα και όλα τα κόμματα ε, για την αλληλεγγύη τους, διότι η αλληλεγγύη μας χρειάζεται να ευχαριστήσουμε και το Συμβούλιο και την Επίτροπο, γιατί ήταν συγκεκριμένη, ήταν ξεκάθαρη. Πρέπει να δείχνουμε ενότητα όποτε υπάρχει διαστρέβλωση της ιστορίας. Παρ' όλα αυτά η συζήτηση δεν έχει χαρακτήρα μόνο ιστορικό, είναι θέμα ασφάλειας, Ελληνική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όσοι πολιτικοί αποδέχονται ολοκληρωτικά καθεστώτα, τότε οι ίδιοι γίνονται συνένοχοι, καταχρώνται της εξουσίας τους επιζημία εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Ένας πολιτικός που ξεχνά την ιστορία, που αποδέχεται τον ολοκληρωτισμό. Δεν θα πρέπει να ονομάζεται Ευρωπαίος. Άρα ενωμένοι και αλληλέγγυοι θα πρέπει να είμαστε. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Λίτκη. Επόμενος μιλητής, ο κύριος Μίλλερ. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν από 30 χρόνια Όταν το Σώμα των Βουλευτών στη Σοβιετική Ένωση καταδίκασαν ε, τη συμφωνία με τον Χίτλερ, που ήταν το τελευταίο που συνέδεσε τους δύο λαούς, φάνηκε να κλείνει αυτό το κεφάλαιο στην ιστορία. Ενώ τώρα φαίνεται ότι ασχολούμαστε εκ νέου με αυτά τα θέματα και προσπαθούμε να αλλάξουμε την ιστορία. Η συμμετοχή της χώρας μου δεν αφισβητείται. Οι Πολωνίδες συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, τους ε, πολέμησαν και υπήρξε ολόκληρο κίνημα κατά αυτών. Έτσι λοιπόν, ότι οι πόνιες γίνονται για το ότι δημιουργήθηκαν ζεστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης με τη δική μας αποδοχή είναι κάτι απαράδεκτο. Ήταν πολύ σημαντικό βέβαια για το Τρίτο Ράιχ η Πολωνία επειδή υπήρχαν πολλοί Εβραίοι. Δεν πρέπει λοιπόν να διαστρεβλώνουμε την ιστορία και τη μνήμη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό πρέπει να το καταδικάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μίλλερ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Νίκολα Μπέρ. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συναδέλφοι. Ως Αντιπρόεδρος είμαι αρμόδιο για το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Σε χώρους σαν αυτούς είναι όλο και σημαντικότερο να μην ξεχνάμε τα μαθήματα της ιστορίας σήμερα, να μην παραμορφώνονται αυτά. Οι στρεβλώσεις ιστορίας δεν λαμβάνουν χώρα μόνο στο ίντερνετ. Ε, Μνημονεύοντα λοιπόν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα σε ένα θέμα που με αφορά ιδιαίτερα, τον αντισημιτισμό παραποιημένη παρουσίαση της ε, εβραϊκής ιστορίας ε, λέει είναι αυτή που οδήγησε ε, στην δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 70 χρόνια μετά υπάρχουν ακόμα θεωρίες συνωμοσία και το κίνημα BDS επιβάλλει μποϊκοτάζ εβραϊκών αγαθών. Αυτό μας θυμίζει γεγονότα τότε που αρνούνταν την ιστορία του Ισραήλ και την ύπαρξή του ε, όπως και η συμπεριφορά ε, στις ψηφοφορίες των Ηνωμένων Εθνών όπου συχνά βλέπουμε αντισημιτισμό να οδηγεί τις πράξεις. Θα πρέπει λοιπόν μαζί ως Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή και ως Συμβούλιο να καταπολεμήσουμε το λόγο μίσους στο διαδίκτυο και να παγιώσουμε τον ορισμό του αντισημιτισμού της International Holocaust Remembrance Alliance. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπέρ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Φέστ, Νίκολας Φέστ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος γνωρίζει λίγο ιστορία ξέρει ότι αυτά που λέει ο Πούτιν ιστορικά είναι λάθος και ότι οι Πολωνοί έχουν κάθε δικαίωμα να κάθονται εδώ. Αλλά ε, δεν είναι, ανήκει εδώ αυτή η συζήτηση. Είναι συζήτηση για τους ιστορικούς. Δεν είναι συζήτηση για πολιτικούς όπως ε, οι πράσινοι και οι αριστεροί πολλοί αυτοί δεν φαίνεται να έχουν ε, ολοκληρώσει επιτυχώς σπουδές ιστορίας Οι πολιτικοί και πολλοί κόσμος δεν, φαίνεται να, δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να συζητά ιστορία Οι πολιτικοί είναι για να οργανώνουν το μέλλον όχι να συζητούν για το παρελθόν Παρότι είναι ενδιαφέρον αυτό και σίγουρα δεν μπορούμε να μιλάμε ε, και να αντιδράμε σε κάθε πρόκληση του Πούτιν και για τις δηλώσεις του να ξεκινάμε εμείς εδώ συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπα, καταλαβαίνω το θυμό των Πολωνών, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ο σωστός ε, τόπος για τέτοιες συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής. Μελμπάρντε, ECR. Ένα λεπτό παρακαλώ, κυρία Μελμπάρντε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι ιστορικός και παρακολουθώ ευχαριστώ τη συζήτηση αυτή. Τον Οκτώβριο το Κρεμλίνο τον Οκτώβριο τότε ασχολήθηκε με την Λετωνία Τελικά κατέληξε να την ελευθερώσει και πάλι. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο επίσης η ιστορία και το σύμφωνο του Χίτλερ είναι κάτι το οποίο δεν συζητιέται αρκετά. Πέρασαν 22 μήνες με τους συμμάχους του Χίτλερ και δεν αναγνωρίστηκε ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν συνυπεύθυνη για τις φρικαλαιότητες Υπάρχουν γεγονότα τα οποία βέβαια δεν ευχαριστούν καθόλου το Κρεμλίνο. Το υλικό για ε, το κίνημα παρτιζάνων στις χώρες της ε, Βαλτικής. Στρεβλώθηκαν όλα αυτά. Κι όμως πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία και να βάζουμε στην πρώτη γραμμή τη μνήμη εκείνων που έχασαν τη ζωή τους και όχι να δοξάζουμε αυτούς που έκαναν τον πόλεμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μελμπάρτε. Επόμενο ομιλητή, η κύριο Σέμ Ντεμιρέλ. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλουμε αλλιόξυνση ούτε ξανά πόλεμο. Εμεί αισθανόμαστε υποχρέωση ω αριστερά. Ωστόσο, οι ρατσιστέ και οι φασίστε ε, απειλούν τη ζωή και ακούμε οι αρχέ ε, πολέμου και δυστυχώς αυτό αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα. Από τη δική μας ιστορία, την ανθρώπινη ιστορία γνωρίζουμε ποια είναι η ορμή του φασισμού, η σκληρότητα ενός παγκόσμιου πολέμου και πόσο σημαντικά, η σημαντική είναι η αντίσταση στο φασισμό. Το Σεπτέμβριο πέρυσι η πλειοψηφία αυτού του κοινοβουλίου θεώρησε ότι είναι το ίδιο πράγμα και ο Χίτλερ και ο Στάλιν. Όταν διαστρεβλώνουμε έτσι την ιστορία, κάθε εναλλακτική πολιτική του καπιταλισμού θεωρείται απολυταρχισμός. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μάθει τίποτα από την ιστορία. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνεχεία τα ίδια λάθη. Όχι, συναδελφοί, ο αγώνας του κόκκινου στρατού μας ε, απελευθέρωση από τη σκοτεινή ιστορία. Όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία δεν μπορεί να αποφασίζει για το μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ευχαριστούμε τον κόκκινο στρατό που μας βοήθησε και τους συμμάχους που σήμερα μας έδωσαν την ελευθερία μας. Η πρόεδρος, ευχαριστούμε. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε το χρονικό όριο για τι αγορές γιατί όλοι θέλουν να μιλήσουν και έχουν πολλά να πουν για το θέμα. Το επόμενο τώρα είναι ο κύριο Κομίν ή Ολιβέρες για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μετά τον ε, πόλεμο γεννήθηκε το ευρωπαϊκό όραμα. Εμείς είμαστε κληρονόμοι και φέρουμε την ευθύνη να συνεχίσουμε να το προωθούμε. Πριν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες είχαν ε, κατησχίσει κατά των ε, δικτατοριών και η ήττα του νατσισμού και του φασισμού ήταν το θεμέλιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς δεν θα γινόταν Είχαμε δημοκρατία, κράτος δικαίου, τις ευρωπαϊκές αξίες, τα ανθρωπινά δικαιώματα, όλα αυτά ήταν τα θεμέλια, όλα αυτά που καταπατούσαν οι δικτατορίε της Ισπανία. Από την άλλη μεριά όμως δεν σε δημοκρατία επί τη ήττα επί του δικτάτορα που πέθανε στο κρεβάτι του, γιατί σήμερα επίσης συνεχίζεται ζωντανή η κληρονομιά του, πολύ ζωντανή. Και ο μετασχηματισμό, ο δημοκρατισμός ε, δεν έγινε όπως σε Ιταλία ή η γερμανια τη δεκαετία του 40 ή όπως έκανε η Πορτογαλία δεκαετία του 70. Σήμερα αυτές είναι εγκαθιδρυμένες στεγανές δημοκρατίες και ξεπέρασαν τον προηγούμενο ολοκληρωτισμό τους. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε για να καταλάβουμε και τις ε, ρίζες αυτής της εκτροπής, αυτής της ολοκληρωτικής εκτροπής που σήμερα έχει πλήξει την Ισπανία θεωρούν ότι για την ενότητα της Ισπανίας θα πρέπει να, να καταπατήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό αφορά και την δικαιοσύνη. Είναι όλα αυτά κληροδοτήματα του φραγκισμού. Ε, είναι ένα ε, ε, εθνικισμός που δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Γκονθάλεθ Πόνς διώκεται από τη δικαιοσύνη ο, ο Και αυτό γιατί έχει κάνει υπεξαίρεση εις βάρος του δημοσίου χρήματος. Θεωρείτε εσείς αγαπητοί μου ότι είναι ολοκληρωτισμός ε, όταν ε, κάποιος ο οποίος είναι φυγόδικος για τέτοια εγκλήματα ε, τώρα να αγορεύει εδώ στο εμικύκλιο δεν, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Έχουμε τώρα 70 χρόνια ε, από τότε που γίνανε πολλά, από τότε που τέλειωσε ο δεύτερο πόλεμο, πόλεμος, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το 1945, δεν τέλειωσε τότε. Τέλειωσε όταν έπεσε το τείχο του Βερολίνου, όταν ο Ερυθρός στρατός αποσύρθηκε από την Ανατολική Ευρώπη. Τότε νικήσαμε τον φασισμό, τον εθνικισμό και τον κομμουνισμό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε γκονσάλε Ο Επόμενο ομιλητή, πρέπει να τον Μπενιφέη. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Για το θέμα τη μνήμη σε αυτή τη θητεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δίνει καλή εικόνα. Το Σεπτέμβριο, κατά τη θέληση τη δική μου ομάδα, αποφάσισατε να ψηφίσετε ένα ψήφισμα, το οποίο τελικά ε, κάποιοι συμπολίτε μας θεωρούν πέραν του κειμένου όχι ως ε, καταδίκη της απολυταρχία, αλλά ως εξίσωση του ναζισμού και μιας άλλης ιστορικής εμπειρίας ε, στην Ευρώπη όσον αφορά την πολιτική που ήταν σοσιαλιστική και κομμουνιστική. Υπάρχει σύγχυση στο κείμενο αυτό. Θεωρείται αθώο το κείμενο όσον αφορά τι συνέπειε, αλλά πολλοί προσβλήθηκαν. Οπότε ζητώ συγγνώμη γιατί εδώ το Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να εκπροσωπήσει την κοινή μνήμη. Να αφήσουμε την ιστορία στους ιστορικούς. Πρέπει να βασιστούμε σε αυτό που ένωσε πραγματικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με καθαρότητα. Στις 25 Οκτωβρίου του 2018 ζητήσαμε καθαρά από τα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν τις νεοφασιστικές, ε, νεοναζιστικές οργανώσεις που ακόμα περηφανεύονται για τις δικτατορίες του παρελθόντος και αντί να κάνουν αυτό θέλω να πω στον συνάδελφο ε, Πάντζα της Λέγκα ότι το Μπέλα Τσάου είναι τραγούδι της αντίστασης όχι μόνο στην Ιταλία, στην Ευρώπη ε, γεννήθηκαμε όλοι χάρη στην αντίσταση που εσείς ε, αμαυρώνετε εδώ πέρα. Θα το πω στα αγγλικά γιατί μπορεί να με ακούσετε. Μιλήσατε τόσο γρήγορα που οι δερμηνεί δεν προλαβαίνουν να σα ακολουθήσουν. Ζητώ συγγνώμη την επόμενη φορά, παρακαλώ λίγο πιο αργά. Ευχαριστώ, ούτω ή άλλω. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Ο κύριο Σιμέτσικα έχει το λόγο τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω πιο αργά, αλλά σλοβακικά, στη γλώσσα μου, μου επιτρέπετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η προσπάθεια των Ρώσων να ξαναγράψει την ιστορία δεν είναι κάτι νέο δυστυχώς συνηθίζεται με την προπαγάνδα που κάνει αυτό που κάνει και όχι μόνο ο Στάλιν. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση όμως και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δυνατόν να σιωπήσουμε απέναντι σε αυτή την προσπάθεια του Πούτιν. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η κοινική συνεργασία μεταξύ δύο καθεστώτων οδήγησε στον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Οπότε, χάρη στη μνήμη των θυμάτων, πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οικοδόμημα αυτό είναι η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δώσει κανείς σε αυτή την φρίκη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε για αυτό το κοινό οικοδόμημα, αλλιώ αυτό θα είναι και το τέλος του. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σιμέτσικα. Επόμενος ομιλητής, Τσόκα. Παρακαλώ. Ναι, να μην διαστρεβλώνουμε την ιστορία, να μην διαστρεβλώνουμε όμως και το παρόν. Και ο κόσμος αναρωτιέται. Αυτή η Ευρώπη, η πολυδάπανη, σε τι έχει αλλάξει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα το, με το 2020. Τίποτα είναι η απάντηση. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ε, γίνονταν οι πόλεμοι με τα τάγκα, με τους... Ε, περάβλους ε, μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των κρατών της Ευρώπης και τώρα έχουμε οικονομικούς, εμπορικούς πολέμους και ρήξει μεταξύ κρατών μελών, διενέξεις που συνεχίζονται ε, όπως και παλιότερα. Βλέπουμε τι γίνεται στη δραματική κατάσταση της ε, Λιβύα, η θέση της Ιταλίας Αφενό, η θέση της Γαλλίας αφετέρου και μια Ευρώπη που δεν κάνει τίποτα. Κάνει τα στραβά μάτια όσον αφορά τον πόλεμο στη Λιβύη. Αν να αποφεύγουμε τους πολέμους ε, για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το να κοιτάμε αλλού δεν είναι η σωστή οδό ε, διαφορές ε, για την επισήμανση των τροφίμων, ε, για διάφορα θέματα και ξαφνικά έρχεται ο πρόεδρος ο πεφωτισμένος Ασόλη που θα σταματήσει να διχάζει τις χώρες, βγάζει τις ε, σημαίες των κρατών που ίδρυσαν αυτή την Ευρώπη από εδώ, από αυτό το κοινοβούλιο. ποιος το πληρώνει όλα αυτά, να υπενθυμίσω κύριε Πρόεδρε, οι λαοί της Ευρώπης, οι χώρες της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αλλά τώρα. Ένα διαδικαστικό έχει ζητήσει ο κύριος Μπουτικόφερ. Παρακαλώ. Έχω μια ερώτηση επί του διαδικαστικού. Επιτρέπεται στο Κοινοβούλιο ένας ομιλητής να λέει ότι μεταξύ του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Επιτρέπεται να λέει τέτοια πράγματα. Επιτρέπεται να τον πούμε τρελό. Ε, στην συζήτηση αυτή δεν δεχόμαστε μπλε κάρτες. Οπότε ήταν αυτό διαδικαστικό ή ήταν μπλε κάρτα. Εδώ σταματάει αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε με τον κατάλογο μιλητών. Και επόμενη μιλήτρια είναι η Ζαμπέλα Έλενα Κλότς. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, οι πρόσφατες προσπάθειες που έχουν γίνει να ξαναγράψουμε την ιστορία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου από πλευρά του κυρίου Πούτιν δεν μας εκπλήσουν. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί. Η Πολωνία, όπως και άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, γνωρίζει γιατί ήταν θύμα όλων των ολοκληρωτισμών και από τις δύο πλευρές που οδήγησαν σε τεράστιες ζημιές και σε πάρα πολλά θύματα. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίζουμε να θυμίζουμε στους φίλους μας στην Ευρώπη ότι ε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ελευθερία και ειρήνη μπορεί να είναι πραγματικότητα ε, μόνο χάρη στις χώρες αυτές οι οποίες απελευθερώθηκαν και από τους δύο ολοκληρωτισμούς και όποιος φλερτάρει με τέτοιου είδους ιδεολογίες πρέπει να βλέπετε σοβαρές συνέπειες. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούν όσοι έχουν σχέσεις με τον Πούτιν. Η προσέγγιση μπορεί να είναι εφικτή μόνο μεταξύ πλευρών που συμφωνούν με τις ίδιες αξίες. Αλλιώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δεν πρέπει να έχουμε πολιτικές σχέσεις που να βασίζονται σε μια πολιτική ιστορία, έτσι όπως τη γράφει ο πρόεδρος της Ρωσίας. Ευχαριστούμε. Σάντρα Περέιρα είναι επόμενη ομιλήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η στρατηγική της δεξιά είναι σαφής. Προσπαθεί να κινητοποιήσει ε, τη μεγαλύτερη πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ξαναγράψει την ιστορία, να προωθήσει τις πιο αντιδραστικές ε, θέσεις. Όμως η ιστορία δεν ξαναγράφεται και ούτε μπορούμε να στρεβλώσουμε την πραγματικότητα. Εδώ δεν υπάρχουν ψέματα ε, που να κρύβουν τα μονοπόλια της σχέσης με το Χίτλερ ε, από χώρες, Γαλλία, Νομέρο Βασίλειο κλπ. Τα ψέματα δεν μπορεί να επιτρέπουν να δημιουργούνται τέτοιες αμφιβολίες για το τι έγινε και τι δεν έγινε. προσπαθούμε να κρύψουμε την πραγματικότητα για να μην συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο προχωράει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος της κυριαρχίας, σε βάρος της δημοκρατίας που σήμερα ε, πλήττονται και είναι και η αιτία της ε, οπισθοχώρησης που διαπιστώνουμε. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, προς την κυρία Περέιρα. Κύριε Κουμπίλιος, έχετε ένα λεπτό. Δεν είναι θέμα η κατανόηση της ιστορίας. Την γνωρίζουμε καλά την ιστορία μας και ξέρουμε επίσης πολύ καλά τι έκανε ο Στάλιν. Σήμερα συζητούμε γιατί μας εκπλήσουν τα όσα κάνει ο κύριος ε, Πούτιν. Ασκεί μία προπαγάνδα στην Σοβιετική παράδοση πήγε για όσα έκανε ο Στάλιν με τον Χίτλερ. Υφιστάμεθα επίθεση προπαγάνδας. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ απλό που πράγμα στον κύριο Πουτίν. Δεν θα τα καταφέρετε αγαπητέ, δεν θα μας διχάσετε για το θέμα αυτό. Εμείς θέλουμε αλήθεια, γιατί η αλήθεια φέρνει ελευθερία. Αυτή είναι η ισχύ της ελευθερίας και της αλήθειας. Θέλουμε το ίδιο για τον ρωσικό λαό. Ελπίζουμε αυτό να πριτανεύσει και στη Ρωσία. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Κουμπίλιος. Μασιμιλιάνο Σμερίλιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε από τους εθνικοσοσιαλιστές για να μπορέσουν να επιβάλλουν μια ρατσιστική, αντισημιστική ε, δικτατορία. Είχαμε ε, το, το ολοκαύτωμα και είχαμε ε, επίθεση προς αυτούς που ήταν εχθροί και πρόκειται για έναν κίνδυνο και είχαμε συνασπισμό διαφόρων δυνάμεων που τελικά κατάφεραν να νικήσουν τον ναζιστή δαίμονα. Οπότε θα πρέπει να δούμε να μην υπάρχει εκμετάλλευση και συγκρίσεις που δεν στέκουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ε, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν στο ολοκαύτωμα και σήμερα έχουμε την ε, άκρα δεξιά που διαδίδει αντισημιτισμό και ρατσισμό. Άρα θα πρέπει η δημοκρατία μας να καταπολεμήσει αυτόν τον κίνδυνο του νέου φασισμού και αυτή η συζήτηση θα πρέπει να είναι αφιερωμένη σε όλους όσοι βασανίστηκαν στο Auschwitz γιατί εκεί στα κρεματόρια ε, γεννήθηκε η αναγκαιότητα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του σοσιαλισμού και του ναζισμού των δαιμόνων της Ευρώπης μας. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε κύριε Σμερίλιο. Κριστιαν Κινέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, θα μιλήσω ρουμάνικα. Εγώ είμαι από τη Ρουμανία και η χώρα μου υπέφερε πολύ από τον φασισμό αλλά και από τον κομμουνισμό. Και εγώ δεν είμαι ευγνώμων στον κόκκινο στρατό, όπω είπαν συναδέλφοι από την αριστερά νωρίτερα. Δεν θέλω να ευχαριστήσω τον κόκκινο στρατό. Ο κόκκινο στρατό κατέκτησε, εισέβαλε στη Ρουμανία, σκότωσε κόσμο, βίασε κόσμο. Ευχαριστώ. Αυτό το κοινοβούλιο ε, πέρασε ένα ψήφισμα το οποίο λέει ότι το σύμφωνο Ρίμπεντροπ Μολοτόφ ε, ήταν μια από τις αιτίες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό αληθεύει. Επέτρεψε στου Ναζί να εισβάλλουν στην Πολωνία και να ξεκινήσουν τον πόλεμο. Ένα κομμάτι της Ρουμανίας ταυτόχρονα είχε ε, κατακτηθεί από τον ε, κόκκινο στρατό. Είναι ένα παρελθόν που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας. Υπήρχαν οι Ναζί στη Γερμανία, αλλά ο Πούτιν λέει ότι ο κομμουνισμός ήταν καταπληκτικός, γι' αυτό είναι παλιάνθρωπος και εγώ θέλω να καταγγείλω ε, την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κινέα. Ο Ζήλ Λεμπρετό, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ε, κατά της Ρωσίας έχει αυτή την επιθυμία να επιτίθεται στη Ρωσία με κάθε μέσο και έτσι ε, ενέψε στον πειρασμό να ξαναγράψει την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στο ψήφισμα τη 19 Σεπτεμβρίου του 2019. Εκεί γράφεται παραθέτω ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε ως συνέπεια άμεση της ε, δυστυχούς ε, συμφώνου μη ε, επίθεσης Ρίμπεντροπ Μόλοτοφ. Σίγουρα υπήρξε αυτό το σύμφωνο και δείχνει τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάζουμε την ε, Σοβιετική Ένωση σε όλη την ιστορία τους και που πρέπει να καταγγείλουμε και εγώ στο Ταλίν. Έχω ποτίσει φόρο τιμής ε, στα χιλιάδες θύματα ε, νους του κομμουνισμού. Αλλά το να λέμε ότι το σύμφωνο αυτό ήταν βασική αιτία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου είναι παραμόρφωση τη ιστορία, διαστρέβλωση τη ιστορία. Εγώ αρνούμε να τη δεχτώ. Α αφήσουμε στου ιστορικού το καθήκον το να ξαναγραφτεί η ιστορία. Η ιστορία αυτή που θα κρίνει άσχημα τη δική μα προσπάθεια χειραγώγηση τη ιστορία. Σας ευχαριστούμε κύριε Λεμπρετόν. Ο Άγγελ Τζαμπάσκη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η Πολωνία ε, είχε δεχτεί την επίθεση ξένων δυνάμεων και είχε διαμελιστεί. Ο Εθνικός Στρατός ε, Άρμια Κραϊόβα προσπάθησε να προσπίσει την ανεξαρτησία της ε, Πολωνίας και θα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής. Αλλά δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να σιωπούμε για τα εγκλήματα των Πολσεβίκων. Θα πρέπει να τα μνημονεύουμε. Είχαμε ένα Βούλγαρο, ονόματι Κρόμα, που προσπάθησε να σώσει 50, περίπου 50 Εβραίους ε, Βουλγαρούς και ε, βομβαρδίστηκε το σπίτι του. Και ότι το υποκομμουνιστική σημαία ε, δίωξε και δολοφόνησε πολλούς ε, Βούλγαρους στη Μακεδονία. Ντροπή στους δράστες αυτών των εγκλημάτων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κιζίλ Γιουρέκ για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν σκοπός μας είναι να διδαχθούμε από το παρελθόν, το πρώτο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι ο εθνικισμός, ε, αλυτρωτισμός, ρατσισμός και φασισμός σημαίνουν πόλεμο. Ο Αδόλφος Χίτλερ με αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία επιδίωξε την πολιτική του. Και ο Αλεκ Κόπεσμαν, ο μεγάλος ιστορικός, ε, δίκιο έχει όταν λέει ότι ο κύριο, οι κύριοι λόγοι για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι δύο λέξεις. Αδόλφος και Χίτλερ. Μερικοί θεωρούν ότι το σύμφωνο Ρίμπετρο Μολότοφ ήταν ο βασικός λόγος του πολέμου και ξεχνούν ότι σχεδόν όλα τα έθνη ε, είχαν συμμετάχει σε μια προσπάθεια κατευνασμού των εντάσσεων. Θα πρέπει να διδαχθούμε από τα παθήματά μας και τα λάθη μας. Θα πρέπει να μάθουμε από τα σφάλματα που έχουμε διαπράξει, να είμαστε κριτικοί απέναντι στην ιστορία μας και να, κατα... και να καταπολεμήσουμε ρατσισμό, αντισημιτισμό. Ε, επίσης, δεν θα πρέπει η ιστορία να είναι προϊόν ιδεολογικοποίησης. Δεν θα πρέπει να ενοχοποιούμε και να δαιμονοποιούμε άλλους για να δημιουργήσουμε τη δική μας ταυτότητα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε κυρίως τον εθνικισμό και να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να συνειδητοποιήσουμε και τις δικές μας σκοτεινές σελίδε της ιστορίας. Σας ευχαριστούμε κυρία Κιζιλ Γιούρεκ. Το λόγο τώρα έχει ο Ραντοσλάβ ε, Σικόρσκι. Ε, φωνές και από την άκρα αριστερά και από την άκρα δεξιά δείχνουν ότι η συζήτηση που ξεκίνησε με την πρωτοβουλία της Πολωνικής Πλατφόρμας των Πολιτών και του PSL είναι πολύ απαραίτητη. Μερικοί ε, εκπλήσονται που ο Πούτιν άλλαξε γνώμη. Από τότε που στο Βεστερπλάτ ε, απέτυσε φόρο τιμής στους Πολωνούς ε, πεσόντες ε, θύματα του Χίτλερ. Και μάλιστα ε, φόρο τιμής και στους Πολωνούς ε, φυλακισμένους και θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τότε δεν κατηγορούσε την Πολωνία. Ε, από την προβοκάσια του Γκλιβίσκη ξεκίνησε ε, και από το Χίτλερ ε, ο πόλεμος. Ερωτούμε λοιπόν γιατί μεταστράφηκε η γνώμη των Ρώσων. Νομίζω ότι ήταν κακή η πολιτική που ακολουθήθηκε τελικά και θα πρέπει να δούμε τι, τι και η σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ολέκας έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και είμαι Λιθουανός. Είμαι από την αριστερά. Αλλά γεννήθηκα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και χαίρομαι που ακούω ότι αριστερά και δεξιά καταδικάζουν τα εγκλήματα αυτά. Στη Λιθουανία Είχαμε 200.000 ε, θύματα Εβραίους ε, συμπολίτε μας. Οι Ναζί, από τους Ναζί. Και εκατοντάδες χιλιάδες ε, ε, εκδιώχθηκαν, πολλοί από αυτούς εκτελέστηκαν. Τα, αρχικά λοιπόν αυτά τα καθεστώτα κόστισαν τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάνε οποιαδήποτε άλλα καθεστώτα. Αν θέλουμε λοιπόν ε, μια δημοκρατική Λιθουανία στην ε, δημοκρατική Ευρώπη, θα πρέπει να τα συζητάμε όλα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν άτομα τα οποία δεν τα γνωρίζουν αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να του ενημερώσουμε για αυτά, για να μπορέσουν να συμβάλλουν στην ελεύθερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βλακά. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Ήγιαψ Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα μιλήσω Γίνονται απόπειρε παραμόρφωση τη ιστορία και αυτό αποτελεί τμήμα μια ευρύτερη στρατηγική ε, στι χώρε τη Βαλτική. Αυτή η προπαγάνδα είναι πραγματικά φρικιαστική. Σε ό,τι αφορά την νομιμοποίηση του ε, Ρίπετροφ Μολότοφ. Θα πρέπει λοιπόν ε, να αμυνθούμε κατά των απόπειρων αυτών. Και σήμερα υπάρχουν κάποια κρατημέλη όπου ακούγονται φωνές ε, λαϊκιστών και αυταρχιστών που κάνουν απόπειρα μια τέτοια προσέγγισης. Δεν ναι. Θέλουμε να αμφισβητήσουμε την ε, πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία. Και μέσα από τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας δίνονται τέτοια παραδείγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιέψ. Επόμενη, Χακαράινεν. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ο κομμουνισμός, ναζισμός, Ισλαμισμός είναι ουσιαστικά μία και αυτή θρησκεία. Εματηρή. Θα πρέπει να μάθουμε στην Ευρώπη ότι Τέτοια στοιχεία δεν πρέπει να τα αφήνουμε να αναδύονται. Κοιτώντα όμως την φιλανδική ιστορία και τον πόλεμο τον οποίο η Φιλανδία έδωσε μόνη της κατά α, του κόκκινου στρατού, του αγαπητού της αριστεράς λόγω της ε, σφαίρας επιρροής μεταξύ Στάλιν και Χίτλερ όπως συμφωνήθηκαν και προφανώς μετά ο Χίτλερ έταξε την ευκαιρία η Φιλανδία αντιστάθηκε